Τη συνεδρίασή μα θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο για την έγκρισή του στην έναρξη τη επόμενη συνόδου. Εάν δεν έχετε καμία αντίρρηση θα διαβιβάσω τα ψηφίσματα τα οποία εγκριθήκανε στους φορείς που αναφέρονται στα οικία ψήφισμα. Η, ε,